Θα καταθέσω και τα ονόματα των όσων επισημένονται μέσα στα κείμενα. Ολοκληρώνεται έτσι αυτή η περίοδος συνόδου. Διακόπτεται. Χαίρετε ε, επόμενη.